Buenos Καλημέρα σας. Να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το νούμερο 13. Περνάμε στο σημείο 13 τη σημερινή διάταξη. Τοποποίηση του κανονισμού 198 του 2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση πολιτικού σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής και για τις ελευτικές δραστηριότητες των αποθεμάτων αυτών. Ο συγγετής είναι ο κύριος Βαλέσα. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την τροποποίηση αυτή και να δώσω το λόγο στον κύριο Βαλέσα. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, δεν προτίθεμαι να εισαγάγω κανένα επαναστατικό σχέδιο για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων της Βαλτικής. Εφόσον μιλούμε για μακροπρόθεσμες προοπτικές, πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον των αποθεμάτων Βακαλάου. Κατά την εκπόνηση της ε, εκθέσεως, θεώρησα ότι χρειάζεται προσαρμογή πρώτα-πρώτα στα προβλεπόμενα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όταν αρχίσαμε να εργαζόμαστε, παντός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ορισμένες αλλαγές για, το, για την ανώτατη βιώσιμη απόδοση, το άρθρο 4, καθώς και το άρθρο 26, την, όπου η αξιολόγηση, μάλλον η περίοδος αξιολογήσεως, αυξήθηκε από 3 σε 4 χρόνια. Εκεί έχουν γίνει ορισμένε αλλαγέ. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να συνεχίσω την μελέτη των αλλαγών και να επανεξετάσω ορισμένα επίμαχα σημεία. Οι αλλαγές που προτείνω είναι απολύτως απαραίτητες, διότι δεν, οι ρυθμίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν συμβαδίζουν πλέον με την κατάσταση των αποθεμάτων βακαλάου στην Βαλτική. Η Κομισιόν είπε ότι θα επανέλθει στο θέμα στην ανάλυση ειδών της ε, Βαλτικής. Ωστόσο, φοβούμε ότι θα σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση. Φαίνεται πως χρειάζεται περισσότερη έρευνα, διότι το θέμα είναι περιπλοκότερο από όσο αναμέναμε και γι' αυτό χρειάζεται συμπλήρωση του υφισταμένου σχεδίου για τα αποθέματα βακαλάου πριν να υποβάλει τη νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι βασισμένη στην επιστημονική έρευνα. Το σχέδιο διαχείρισης το ίδιο θεωρώ ότι είναι εντάξει. Βρίσκει ότι η κατάσταση των αποθεμάτων Βακαλάου είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πιστευόταν. Δεν είναι όμως αρκετά ευέλικτο το σχέδιο διαχείρισης. Οι ψαράδες μας λένε ότι τα αποθέματα ε, βακαλάου στην Βαλτική είναι σε καλή υγεία. Τα προηγούμενα χρόνια οι επιστήμονες είχαν πει ότι σε τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να αυξηθούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα λίευματα και κατά 40%. Ωστόσο, οι ποσοστώσεις έχουν μπλοκαριστεί για την ώρα σε επίπεδο που δεν είναι ενδεδειγμένο. Και προβλέπεται μονάχα 15% αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι στο ανατολικό τμήμα της ε, θάλασσας αυτής υπάρχει τόσο απόθεμα ώστε η κατάσταση του είδους είναι πολύ χειρότερη και έχουν, ε, συμβεί και, ε, έχουν σημειωθεί και περιπτώσεις κανιβαλισμού των ψαριών. Προτείνεται μάλιστα μείωση για το 2013 των ε, αλλιευμάτων. Έτσι νομίζω, αναμένοντας την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε κάποιες αλλαγές που να καταστήσουν πιο εύκαμπτο το μηχανισμό της ρύθμισης των ε, ανώτατων ε, αλλιευμάτων. Αλλά χρειαζόμαστε και ορισμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, τον κίνδυνο κανιβαλισμού. Ε, χρειαζόμαστε κάποιε ενδείξει σχετικά. Οι προτάσει μου, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε ευχολόγια. Εγώ επιθυμώ οι προτάσεις που θα κάνω να βασίζονται σε επαληθευμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Και γι' αυτό μελετώ μια αλλαγή που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο εύκαμπτοι σε ό,τι αφορά τα ΤΑΚ. Βέβαια, όπως είπα, πάντοτε στην βάση επαληθεύσιμων επιστημονικών δεδομένων. Εξετάζουμε τώρα, όπως είπα, το ανατολικό απόθεμα που είναι και το μεγαλύτερο. Αλλά θα πρέπει να εγκύψουμε και στην περίπτωση του δυτικού αποθέματος και μάλιστα σύντομα. Και εδώ ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει υπόψη μας τα σχόλιά της για το δυτικό απόθεμα του Βακαλάου στην Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο της Κομισιόν, παρακαλώ έχετε το λόγο. Μάλλον όχι. Καταρχήν ε, να δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή. No, Κανένας ε, δεν υπάρχει να παρέμβει εδώ. Bueno, pues parece que no, la Comisión... Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της Επιτροπής. Παρακαλώ, κύριε Κούν. Oh, Ευχαριστώ. Βεβαίω δεν πρόκειται να εκπροσωπήσω την Κομισιόν. Ήδη οι εμπειρίες του κυρίου Βαλέσα που περιλαμβάνει στην έκθεσή του για το πολιετές σχέδιο διαχείρισης τις υποστηρίζω Καφέ παρακαλώ. Αλλά εδώ ο άνθρωπος που φέρνει το καφέ μου λέει δεν είναι καφέ, είναι απλώς μαύρο ζούμι. Η Κομισιόν δεν είναι παρούσα. Αυτό νομίζω δείχνει, σήμερα δηλαδή, δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα του Βακαλάου στην ε, Βαλτική τα πήγανε καλά σε συνεργασία με τους ντόπιου ψαράδες αλλά και με τους επιστήμονες και με τα ΡΑΚ, τα Περιφερειακά αριστικά Συμβούλια. Πριν από λίγα χρόνια η κατάσταση του αποθέματος ήταν, σε πάρα πολύ άσχημη. ήταν πάρα πολύ Ο κύριος Βαλέσα τα γνωρίζει αυτά. Και οι Γερμανοί ψαράδες αλλά και οι Πολωνοί και οι, από τις βαλτικές χώρες φοβούνταν ότι στο μέλλον δεν θα είναι πια το ψάρι αυτό από εκείνα που αλλιεύονται σε μεγάλους αριθμούς. Λήφθηκαν διάφορα μέτρα και το απόθεμα αυξήθηκε αλματοδός. Εδώ προστίθενται βέβαια και κάποιες φυσικές εξελίξεις, δηλαδή κάθε 10 χρόνια περίπου μπαίνει η ποσότητα αλμυρού νερού από άλλη θάλασσα στη Βαλτική και αυτό ενισχύει την τάση γονιμοποίησης του ψαριού. Πρέπει να φροντίσουμε να διατηρηθεί στα σωστά επίπεδα το απόθεμα. Ο Βαλέσα σωστά είπε, όχι, θέλουμε, όχι θέλουμε μονάχα την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η βιομάζα του ψαριού αυτού δεν, πρέπει, δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ας πούμε μάζα. Οι επιστήμονες ε, έχουν ε, υπολογίσει ότι θα πρέπει να είναι περίπου στις τάξεις των 200.000 τόνων. Διότι τότε, ε, αν ξεπεραστεί το όριο αυτό, και ε, κανιβαλιστικά επεισόδια μπορεί να τύχουν, αλλά ε, υφίσταται το πλήγμα και νεαρές ρέγγες, νεαρά σκουμπριά κτλ. Γιατί ο βακαλάος είναι αρπακτικό ψάρι. Χρειάζεται λοιπόν μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση. Τα, τον τελευταίο καιρό ακούμε και άσχημες ειδήσει. Ότι η τιμή του ψαριού αυτού στη Βαλτική έχει πέσει πολύ. 68 λεπτά του ευρώ ανά κιλό. Και μάλιστα και 70 τόνοι πήγανε για ηχθιάλευρα. Προσοχή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ακούσουμε από την Κομισιόν άποψη για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την διατήρηση της συνολικής ισορροπίας των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων στην Βαλτική. Μαζί με συνεργασία βέβαια με τις χώρες μέλη, με την επιστημονική έρευνα, διότι χρειαζόμαστε βέβαια πολύ περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να δούμε πώς ε, θα εξελιχθεί Αυτά, αυτές τις ε, παρατηρήσεις είχα να κάνω. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λουβίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Μια πρώτη σκέψη που κάναμε χθε. Ε, ο κύριος ε, Οντόνικ ήταν εδώ από το Πελαγικό Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβουλίο και μίλησε για το απόθεμα του Σαφριδιού και ήταν σαφής ότι το πελαγικό ρακ στα βορειοδυτικά ύδατα ήθελε μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Θέλει να μπορεί να σχεδιάσει ε, επί των ελευμάτων ε, μακροπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν ε, βρισκόμαστε τώρα σε μία σύγκρουση με το Συμβούλιο και το Συμβούλιο θέλει ε, ετησίω να εφαρμόσει το FMSY, τότε οι διακυμάνσει για τον κλάδο θα είναι ιδιαίτερα ζημιογόνε. Ναι, και αυτό θα σημαίνει συν 23% ε, πριν δύο χρόνια και συν 30% πέρσι. Όμω δεν του αρέσουν αυτέ οι διακυμάνσει, γιατί ετησίω πρέπει να γίνονται αλλαγέ στον κλάδο και δεν ξέρουν ποιο θα είναι το εισόδημα. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κλάδος ε, επί της ουσίας υποστηρίζει να έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης χωρίς μεγάλες διακυμάνσει. Αυτό έχουμε σήμερα στη Βαλτική και εγώ υποστηρίζω την προσέγγιση αυτή. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αυξάνουμε ή να μειώνουμε ε, τα αλλιεύματα πάνω ή κάτω του 15%. Αυτό έχει να κάνει και με την αρχή της πρόληψης. Και είπατε ότι ο κάδος της Βαλτικής έχει ανακάμψει. Και αυτό ήταν και το μήνυμα του ISIS τα τελευταία δύο-τρία έτη, αλλά και πάλι φέτος μας είπαν και πάλι πρέπει να μειώσουμε. Και ακόμη και αν έχουμε εφαρμόσει το συμπλήν 15% και αφήσαμε ε, κάποια δυνατότητα για λανθασμένους υπολογισμούς, είναι πολύ σημαντικό να εμείνουμε στην αρχή αυτή, και να μην, αυξάνουμε, να μην τις 40% γιατί το ISIS ε, θα μας λέει κάτι το ένα έτος και μετά το επόμενο έτος θα μας λένε όχι, όχι, κάναμε λάθος, πρέπει να μειώσουμε 55% γιατί αυτή η κατάσταση ήταν δεκαετία του 90 και δεν πρέπει να την επαναλάβουμε κατά τη γνώμη μου. Είναι λοιπόν σημαντικό να εμείνουμε στην αρχή αυτή. Τώρα για τον κανιβαλισμό. Αναφέρετε τον κανιβαλισμό, αν δείτε την έκθεση ISIS, του Συμβουλίου για τη Διερεύνηση τη ε, θάλασσα. Ε, υπάρχει μία έκθεση για το περιεχόμενο του στομάχου του γάδου ε, και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ περιθωριακό και είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό του κανιβαλισμού, το 92 ε, ξεκίνησε αυτή η φήμη για μεγάλο κανιβαλισμό, όμως αν δείτε τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πολύ χαμηλό περιεχόμενο στο στομάχι του γάδου. Ε, έτσι λοιπόν δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, δεν πρέπει να λέμε ότι ο γάδος, τα, τα ψάρια θα φάνε το ένα το άλλο αλλά είναι ε, το κύριο απόθεμα στη Βαλτική θάλασσα και πρέπει να διατηρήσουμε γη τη Βαλτική θάλασσα. Αν δείτε λοιπόν το απόθεμα του γάδου ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο τη δεκαετία του 1980 και είχαμε γάδο και μέχρι τον κόλπο της Βουτογιάς. ενώ τώρα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Βαλτικής, στα πολωνικά ύδατα κυρίως, και αυτό σημαίνει ότι οι Σουηδοί παραπονιούνται οι Σουηδοί Ελλείς ότι δεν φτάνει ο γάδος ε, καν τις Σουηδικές ακτές, δεν ανεβαίνει η βόρεια στον κόλπο όπως είχαμε τη δεκαετία του 80. Η Βαλτική λοιπόν έχει την ικανότητα να παράγει πολύ περισσότερο γάδο σχέση με το τι παράγει σήμερα και χάρη του οικοσυστήματος θα έπρεπε να επιτρέψουμε την αύξηση του αποθέματος ε, και όχι να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή την μετριοπαθή αύξηση που είδαμε τα τελευταία έτη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαλέση, θέλετε να απαντήσετε. Α, μάλιστα, έχουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank uh, you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που αργοπόρησα και δεν παρακολούθησα εξ αρχής τη συζήτηση. Θα ήθελα να διχοτομήσω τη συζήτηση. Πρώτον, η ευθυγράμμιση που προετοιμάσαμε πρόκειται για μια τεχνική τροποποίηση του κανονισμού περί πολιετού σχεδίου διαχείρισης του γάδου. Σε αυτό το στάδιο θεωρούμε ότι πρόκειται για μία νομικού χαρακτήρα άσκηση. Δηλαδή, προετοιμάσαμε τον κανονισμό για να τον ευθυγραμμίσουμε ως προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, το δεύτερο τμήμα, μελλοντικό σχεδιασμός. Ο γενικός μου διευθυντής, αν δεν απατώμε, ήταν εδώ στην Επιτροπή Αλληλείας και είπε την περασμένη φορά ότι συνεργαζόμαστε με τους επιστήμονες για την εκπόνηση νέου σχεδίου που θα καλύπτει το κομμάτι των ε, ψαριών, των πελαγικών ειδών, των αποθεμάτων ε, γάδου στα πλαίσια του γενικότερου οικοσυστήματος στη Βαλτική. Υπάρχουν και άλλοι συντελεστές όμως που περιορίζουν την κατανομή του αποθέματος. Πολύ σε εντελεστές οικολογικού χαρακτήρα στη Βαλτική. Γιατί είναι φάλμηρο το νερό δίπλα στη Βαλτική και αυτό και άλλοι συντελεστέ περιορίζουν την ισότιμη κατανομή του αποθέματος. Από τη Βόρεια Θάλασσα εισέρχονται και αλμυρά ύδατα και πρόκειται δηλαδή για μια σειρά αιτιών ε, που οφείλονται στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Μου μιλήσατε επίσης για το 40% της ευελιξίας. Είδαμε αυτές τις ε, βαθιές αλλαγές ε, που σημειώθηκαν στον τομέα και τι επιπτώσει είχαν στον κλάδο. Όλοι θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερη κατάσταση αν σημειωθεί αύξηση. Τι γίνεται όμως με τη μείωση, διότι αυτό ήταν ένα καλό δίχτυ ασφαλείας ε, και για τους αλληλείς ε, και για τον κλάδο όταν γίνονται ε, μικρές αυξήσεις γιατί και οι μειώσεις περιορίζονται στο 15% με τα πελαγικά είδη χρειάστηκε να μειώσουμε κατά πολύ τα ετήσια τάκ και φυσικά έτσι είχαμε καλά αποτελέσματα για το απόθεμα και φέτος και για το μέλλον. Με αυτές Αυτές οι μεγάλες μειώσεις είναι επώδυνες πάντοτε και γι' αυτό προτείνουμε 15-20% μόνο ευελιξία σε αυτό το πολιετές σχέδιο διαχείρισης για τα ΤΑΚ. Αυτή είναι η ευελιξία που δίνουμε για τα ΤΑΚ σε αιτήσια βάση. Λάβαμε και νέες επιστημονικές συμβουλές και βλέπετε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά αποθέματα στη Βαλτική. Το δυτικό απόθεμα όπου παρατηρήθηκαν διαφορές σε σχέση με τον προσδιορισμό του συντελεστή της εθνισιμότητας των ψαριών στα πλαίσια του σχεδίου διαχείρισης του γάδου. Στα πλαίσια του νέου σχεδίου θα επανεξετάσουμε αυτά τα στοιχεία και όπως σας είπα, επεξεργάζονται το σχέδιο επιστήμονες, το ίδιο και οι υπηρεσίες μας σε συνδυασμό με το Συμβούλιο που θα καταρτήσει και την ανάλυση αντικτύπου. Συμβουλευτήκαμε και το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο πέρα από τους επιστήμονες και τον Ιούλιο έχουμε προβλέψει ήδη σύσκεψη με τους ενδιαφερόμενους και τα κράτη-μέλη για το απόθεμα αυτό και πάλι δηλαδή για να συζητήσουμε πώς θα προχωρήσουμε με το σχέδιο διαχείρισης για πολλά είδη. Μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις ε, θα εκπονήσουμε τη νέα πρόταση. Όμως, ως προς τις τεχνικές ε, τροποποιήσεις, θα σας συμβούλευα να ακολουθήσετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Eh, Βαλέσα. Ευχαριστώ για τα σχόλια των ε, συναδέλφων. Έχω το εξής να πω. Πρόκειται για την στάνταρτη διαδικασία ευθυγράμμισης με τα προβλεπόμενα από την ε, Συνδίκη της Λισαβόνας. Εκεί την τροποποίησε την διαδικασία αυτή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι και εμείς μπορούμε εδώ στην Επιτροπή Ελίας να εισαγάγουμε ορισμένες τροπολογίες σχετικά εφόσον βασίζονται βέβαια σε επιστημονικές ε, εκτιμήσεις. Και ακόμα κάτι σχετικά με τις ε, επιστημονικές σύμβουλες. Ακόμα και αν εξετάσουμε το τι λένε οι ίδιες επιστημονικές οργανώσεις, βλέπουμε ότι οι συμβουλές τους αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Αυτό οφείλεται και στο ότι αλλάζουν και οι μέθοδοι διεξαγωγής των ερευνών τους. Γι' αυτό και έχει αναβληθεί μέχρι τώρα η εφαρμογή του ε, σχεδίου διαχειρίσεως και κατ' επανάληψη μάλιστα των αποθεμάτων της Βαλτικής. Χρειάζεται λοιπόν να ζητήσουμε συμβουλές από περισσότερους οργανισμούς. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε μερικές μόνο απόψεις και γι' αυτό επιμένω. Χρειάζεται λοιπόν να ακούσουμε τις επιστημονικές συμβουλές, αλλά να έχουμε πλείονε πηγές επιστημονικών ε, συμβουλών, όχι μόνο χαμία. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Και χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ας περάσουμε σημείο 15 της ημερησίας διάταξης, λέει ο Πρόεδρος. Πρόταση κανονισμού Δρομοποίηση του κανονισμού 2371 για τη διατηρήση και βιώσιμη των λευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτική. πολιτικής. Ξέρετε ότι η προθεσμία λύγει στα τέλη του έτους, δεν θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης γιατί δεν θα έχουμε τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΛΠ να έχει εγκριθεί πριν από αυτή την ημερομηνία. Έτσι λοιπόν έχουμε στενό χρονοδιάγραμμα αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε την παράταση πριν να ολοκληρωθεί το έτος. Η Κομισιόν έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει την πρόταση κανονισμού. Good morning. Uh, Καλημέρα. Όντως, θα θέλαμε να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα σε σχέση με την όλη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Ε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβετε ποιο είναι το πλαίσιο. Είναι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα για αυτό το άρθρο δηλαδή που εισαγάγαμε στην κοινή αλληλευτική πολιτική και ήταν, ε, υπήρχε και πριν το εισάγουμε γιατί το 70 άρχισε να ισχύει με κάπως διαφορετικούς όρους αλλά τότε άρχισε ε, από ε, τα έξι κράτη μετά τα δέκα και στη συνέχεια συνέχισε να ισχύει για να προστατευθούν οι στόλοι, κυρίως οι μικροί αλληλευτικοί στόλοι, επιτρέποντας τα κράτη-μέλη να αποκλείσουν σκάφη από άλλα κράτη-μέλη στην τότε ζώνη των 6 μιλίων που έγινε 12 μιλίων. Και έτσι, μπορέσαμε να κατοχυρώσουμε τις σχέσεις των ε, των γειτονικών χωρών, γιατί σας μίλησα για τη ζώνη των 6 και στη συνέχεια 12 μιλίων. Το 83 όταν έγινε η πρώτη συνολική, το πω έτσι, μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, ε, επανεισάγαμε τη διάταξη και δεν άλλαξε τίποτε έκτοτε εκτός από μια προσωρινή απόκληση προς την ελεύθερη πρόσβαση. Ε, διότι έτσι αποκλείονται από την ελεύθερη πρόσβαση κάποια σκάφη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε αποφάσισε ότι ε, θα λαμβάναμε νέα απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα με κάθε ένα διαπραγμάτευση. Τώρα λοιπόν που τροποποιούμε το βασικό κανονισμό, προτείνουμε και πάλι προσωρινή απόκληση, πάλι δεκαετούς ε, διάρκειας ε, μέχρι το 2022. Ξέρετε ότι έχουμε καθυστερήσει ε, με την έγκριση του νέου βασικού κανονισμού, αλλά έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να καλύψουμε αυτό το νομικό κενό προτείνοντας μια προσωρινή διετή παράταση ισχύω της ίδιας ε, διάταξη, όπως βλέπετε στο άρθρο 17.2 του βασικού κανονισμού, δεν τροποποίησαμε τη διατύπωση. Επαναλαμβάνουμε την αρχή της, του αποκλεισμού της πρόσβασης στη ζώνη των 12 μιλίων, όπως και πριν. Άδεια πρόσβαση όπως έχουμε στο παράρτημα 1 του βασικού κανονισμού παραμένει και επίσης οι σχέσεις γειτονίας όπως έχουν θεσπιστεί παραμένουν. Προτείνουμε διετή παράταση διότι θεωρούμε ότι επαρκεί ο χρόνος ε, για την έγκριση του νέου βασικού κανονισμού. Με το που εγκριθεί ο νέος βασικός κανονισμός, θα ακυρωθεί ο ισχύοντας κανονισμό, ο ισχύον κανονισμός και στην ε, συνέχεια όπως σας είπα θα έχουμε μια δεκαετή παράταση από το 2012 έως το 2022. Δεν αλλάζουμε τίποτα, προτείνουμε διετή παράταση όπως σας είπα ήδη και κινούμαστε στο πλαίσιο της ε, τροποποίησης του βασικού κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάντωνος, συζητητής, έχει το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τη σαφή εξήγηση σε σχέση με το που βρισκόμαστε. Και τι έκπληξη η νέα μεταρρύθμιση δεν θα είναι έτοιμη εγκαίρως. Αυτό ήταν και σαφές ήδη πριν να γνωρίζουμε ότι είχαμε τόσες πολλές τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό επιβεβαίωσε κάτι που γνώριζαμε όλοι εδώ και κάποιο καιρό, ότι δεν θα είναι έτοιμη η μεταρρύθμιση κίνηση ελευθερικής πολιτικής εγκαίρω. Είναι ενδιαφέρον ότι το Συμβούλιο μαζί της επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί Από ό,τι φαίνεται δεν θα τα καταφέρουν μέχρι τα τέλη του έτους και υπάρχουν λόγοι να συμφωνήσουμε με αυτό, όμως και εμείς ζητήσαμε ε, κάποιο χρόνο να κινηθούν και αυτοί κάπως πιο γρήγορα σε σχέση με τα σχέδια διαχείρισης. Και ίσως ε, μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατή ανταλλαγή, αυτό το παζάρι. Κατά την άποψή μου, Υπάρχουν ε, πάρα πολλά θέματα, πολλά τμήματα της μεταρρυθμιστικής ελευθερικής πολιτικής μπορεί να θεωρήσει ότι ε, είναι ευρωϊκά, όμως όπως φαίνεται από την πρόταση της Κομισιόν αυτός είναι ένας τομέας όπου έχει γίνει αξιολόγηση, ή επαναξιολόγηση και έχει γίνει αποδεκτό ότι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από τα κράτη-μέλη έχουν ε, μειώσει την πίεση στις πιο ευαίσθητες βιολογικά περιοχές και έχουν ε, συνεισφέρει ε, στο να υποστηριχθεί η μικρή αλευτική δραστηριότητα, η ρεσταχνική αλευτική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε ένα τέτοιο κανονισμό και όταν αναφερήσαμε για τελευταία φορά την κοινή ελευτική πολιτική, το 2002 εγώ ψήφισα υπέρ μεταρρυθμίσεων που θα επέκτηναν ε, και την απόσταση πέρα από τα 12 μίλια και θα καθιστούσαν αυτό το καθεστώς μόνιμο. Και εξακολουθώ να επιθυμώ να θετεθούν σε εφαρμογή αυτές οι αρχές. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να καθυστερούμε με κάτι προσωρινό που θα διαρκέσει δεκαετή, γιατί δεν δημιουργούμε ένα μόνιμο καθεστώς και να έχουμε κάποιες ε, αναθεωρήσεις ή κάποιο έλεγχο σχετικά με την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος. Όπως και να έχει, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό να αφήσουμε το καθεστώς αυτό να λήξει αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν με την ιδέα να επεκταθεί, τουλάχιστον να παραταθεί μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2014. Και όταν θα έρθει η νέα μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΛΠ, θα το επιλύσει αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν κάποια σχόλια να κάνουν στο στάδιο αυτό πριν ε, να εκπονηθεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Κύριος Ντέιβις. Έχω μπερδευτεί λίγο από αυτά που είπε ο Ιαν, διότι πρώτα προκάλεσε την προσοχή μου λέγοντας ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για να μπει κάποια κίνηση στα πολιετή σχέδια του Συμβουλίου. Μετά μίλησε για μια παράταση δύο ετών. Ας ρωτήσω την Επιτροπή, ποιε είναι οι νομικές επιπτώσεις της καθυστέρηση αυτού του νομοθετήματος. Μπορεί να χρησιμεύσει ως μοχλός, διότι κάτι χρειάζεται για να... Κάποιος μοχλός χρειάζεται για να φέρουμε το Συμβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άλλο κανεί, η κυρία Φράγα. Δεν θα τοποθετηθώ σε σχέση ε, με την παράταση του χρόνου προ την Κομισιόν, αλλά εγώ συμφωνώ όμως είπε ο συγητής. Καταρχήν, ε, δεν συμφωνώ αυτή η παρέκκληση να είναι μόνιμη, είναι μία παρέκκληση γενική, την υποστηρίζουμε και δεύτερον, ούτε συμφωνώ η αιτιολόγηση να είναι ότι μέσα στα 12 μίλια τα κράτη-μέλη έχουν μειώσει την ελευτική πίεση. Κανένα δεν υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Αν διατηρηθεί λοιπόν θα είναι για άλλους λόγους, όχι για αυτούς που ανέφερε ο εισηγητής. Εγώ δεν συμφωνώ με το σκεπτικό του, αλλά τέλος πάντων θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η παρέκκληση μέχρι να επιληθεί το θέμα του βασικού κανονισμού. Κύριε Χάτον. Ευχαριστώ. Απαντώ στην κυρία Φράγα. Είπα ότι δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην γίνει μόνιμο το μέτρο. Μόνιμο χαρακτηριστικό είπε στην ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η προκατοχή μας έκαναν κάποιο σχέδιο διαχείρισης και πριν από την κοινή αλληλευτική πολιτική. τονίζω τα σχόλια που βρίσκει αντιφατικά η κυρία Φράγα σε σχέση με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> σχετικά με την οικονομική σταθερότητα και τη μείωση της πίεσης στα αλλιεύματα στις περιοχές αυτές. Έχω βεβαίω απόψει, αλλά το μόνο που έκανα δεν ήταν να προβάλλω τι απόψει μου, αλλά να διαβάζω το τι έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, λέει ο πρόεδρος της Κομισιόν, να μην επισέλθω σε θέματα τακτική των διαπραγματεύσεων μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Να απαντήσω τον κύριο Ντέιβις όμως. Αν δεν εγκρίνεται τη νομοθεσία πριν τέλους του έτους, η μόνη σημαντική βέβαια επίπτωση είναι ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και δεν θα ισχύει πλέον το παράδειγμα 1 της ρύθμισης. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή πλέον διμερείς ρυθμίσεις για την πρόσβαση. Οπότε θα υπάρχει πλήρης ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα ύδατα της Ένωσης. Αυτή είναι η νομική επίπτωση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την ύπαρξη των πολυετών σχεδίων διότι όπου υπάρχουν τέτοια καλύπτουν και τις ζώνες 12 μιλίων, δεν διασυνδέονται, ξαναλέω, δεν μπαίνω σε θέματα τακτικής και πολιτικής των ε, θεσμικών οργάνων, αλλά θα έχουμε full free access regime, χωρίς δυνατότητα των χωρών μελών να περιορίζουν την, το δικαίωμα μόνο στα δικά τους ε, σκάφη. Για τις περισσότερες χώρες μέλη νομίζω θα αποτελέσει πραγματικό σοκ Αυτά είναι τα γεγονότα ωστόσο. Άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι δεν νομίζω να είπα ότι πρόκειται για μόνιμο χαρακτηριστικά της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είπα ότι ήταν χαρακτηριστικό και πριν από την αλληλευτική πολιτική. Και κάθε φορά που το αξιολογήσαμε, προτείναμε παράταση, ναι. Και κάθε φορά που προτείναμε την παράταση, το Συμβούλιο τότε που ήταν ο μοναδικός νομοθέτης, τότε λέω, το δέχτηκε, τη δέχτηκε την παράταση. Όπως είπε και η κυρία Φράγα βέβαια, υπάρχουν δύο ξεκάθαρες πτυχές εν προκειμένου. Αφενός πρόκειται για απόκληση από την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης. Έχουμε κάνει και επιστημονικές ας πούμε, μελέτες που μας οδηγούν να πούμε ότι δεν βλέπουμε λόγο να ξεφύγουμε περισσότερο από την ελεύθερη πρόσβαση όπως είπα πάντοτε το σχέδιο αυτό, πάντοτε το χαρακτηριστικό αυτό ήταν προσωρινό, αλλά και πάντα ζητήσαμε την παράταση. Και θεωρούμε ότι πρέπει κάπου κάπου να επανεξετάζουμε τις ε, ρυθμίσεις που προκύπτουν από πολύ σημαντικές διατάξεις της συνθήκης. Και γι' αυτό και στην ε, πρότασή μας για την κοινή αντιευτική πολιτική, και άλλα και τώρα το ξαναπροτείνουμε. Ο κ. Χάντον πρότεινε και την επέκταση στα 12 μίλια. Να το συζητήσουμε. Ίσως να γνωρίζετε την στάση μας από πριν. Υπάρχει ωστόσο ένα πράγμα και θα επανέλθω στο αρχικό μου σχόλιο. Μπορείτε να διαπραγματευτείτε πολύ και εμείς θα συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις. Αν όμως δεν εγκριθεί ο κανονισμός πριν από το τέλος του χρόνου και μάλιστα να αρχίσει να ισχύει κιόλας, ξαναπερνούμε στο σύστημα της ε, ελεύθερης πρόσβασης και νομίζω ότι κανείς δεν θα θέλει κάτι τέτοιο, καμιά χώρα μέλος δηλαδή. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Αν όμως θέλετε, ευχαρίστω να επιχειρηματολογήσουμε γιατί εμένουμε σε αυτά τα οποία διαθέτουμε ήδη. Θα αρκεστώ σε αυτά τα σχόλια. Ο κ. Ε, εγώ υποστηρίζω απολύτω τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πρόκειται για αρχές οι οποίες έχουν αποδείξει την αξία τους και οφείλουν να συνεχίζουν. Αυτό είπε άλλωστε και πριν η κυρία Φράγα. Έχουμε αυτή την ζώνη προστασίας της αλίας των 12 μιλίων μέσα στα πλαίσια της Ένωσης με διμερείς συμφωνίες. Η ρύθμιση που έχει γίνει είναι ότι μέσα σε αυτή τη ζώνη προστασίας μπορεί μέσα σε μια μικρότερη ζώνη των τριών μιλίων να αλλιεύουν και άλλα σκάφη. Και αυτό, αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλά και θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν βλέπω κανένα λόγο να ε, επιφέρουμε ιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες μόνο σύγχυση θα προκαλέσουν και μόνο νέα προβλήματα θα φέρουν. Γι' αυτό, προτείνω, ε, γι αυτό μάλλον υποστηρίζω τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ντέιβις. ως πραγματικό εργαλείο για τα πολιετή σχέδια. Αυτό θα είναι σαν ένα ε, όπλο για την ε, ε δευτέρα παρουσία για τη μέρα των κατεραμένων, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια άλλη εναλλακτική. Μάλιστα. Να περάσουμε στο σημείο 16 για το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης ε, Γρυλανδίας. Ε, ξέρετε ότι στις 2 Φεβρουαρίου του 2012 ε, ισχύει αυτό το πρωτόκολλο για μια περίοδο τριών χρόνων από την 1η Ιουλίου του 2013. Το Συμβούλιο πρέπει να μας στείλει το επίσημο αίτημα έγκρισης κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και εδώ το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ή όχι. Καταρχήν θα έχουμε μία παρουσίαση από την πλευρά της Κομισιόν. Που δεν είναι εδώ. Δεν θα έρθει η Κομισιόν καν να παρουσιάσει το πρωτόκολλο. Έχουμε έναν εισηγητή, τον κύριο Κρίστενσεν. Αλλά αφού δεν είναι δε Κομισιόν, μάλλον ε, δεν θα απευθυνθείτε Κομισιόν όμω, ε, θέλουμε να στείλουμε ένα επίσημο παράπονο μέσω των εκπροσώπων τη Κομισιόν που είναι εδώ σήμερα. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει τουλάχιστον να σέβεται κατά το ελάχιστο αυτή την Επιτροπή και όταν ε, παρουσιάζουν ε, οι εκπρόσωποι τη Κομισιόν πρέπει να παρευρίσκονται εδώ διαφορετικά. Δεν σέβεστε καθόλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε να σα το γνωστοποιήσουμε αυτό. Ε, τώρα βέβαια είναι σαν να κατηγορούμε αυτού που βρίσκονται εδώ, αλλά κοιτάξτε όσου αποσιάζουν τι να πω αφού δεν είναι εδώ. Κύριε Κρίστενσεν. Δεν ε, υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος ε, να συζητήσουμε. Έχω μόνο τέσσερις ερωτήσεις που ήθελα να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τις στείλω λοιπόν γραπτός, ελπίζω ότι θα λάβω απάντηση. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσω την έκθεσή μου. Ευχαριστούμε κυρία Λαβίνη τώρα. Συμφωνώ με σας Πρόεδρε. Έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο δείχνει αυτό και ότι αν, στείλουμε, αν στείλει ο κύριος Κρίστασεν γραπτό στις ερωτήσεις, πάει να πει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν ε, λαμβάνουν γνώση τα μέλη της Επιτροπής των ερωτήσεων. Τι να πω, ας εγγραφεί το σημείο στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης για να ακούσουμε κι εμείς, ε, να μάθουμε ε, για το περιεχόμενο των συζητήσεων του κυρίου Κρίνθας με την Επιτροπή. Κυρία Φράγκο. Δεν ξέρω αν θα αναβληθεί η συζήτηση. Εγώ είχα μια σειρά ερωτήσεων βέβαια, αλλά τι να κάνω, να τις κρατήσω για την επόμενη φορά. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να το θέσουμε στην μερική διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας. Πάντω, αν κάποιο θέλει να στείλει κάποια ερώτηση γραπτό, ευχαριστώ να τη διαβάσουμε, να τη στείλουμε. Μου λένε ότι θα έρθουν σε πέντε λεπτά. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί καθυστερούν. Να συνεχίσουμε εμείς με τη συνεδρίασή μας. Και φυσικά θα στείλουμε και αυτή τη διαμαρτυρία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα παραπονηθούμε. Για τα διάφορα. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι. Απλώς να σας πω ότι στον τριμερή διάλογο ο κ. Γκάλεκερ δεν είναι εδώ. Το αποτέλεσμα για τα εμπορικά μέτρα είναι το εξή. Καταλήξαμε χθε σε μια συμφωνία και νομίζω ότι ολοκληρώνεται το θέμα αυτό. Τώρα, για το συστάσεις που εγκρίθηκαν τους συντονιστές, ε, έχετε λάβει το σχετικό έγγραφο και θεωρείτε ότι εγκρίνονται αν δεν ε, έχετε αντίρρηση. 11 Ιουλίου θα συνεδριάσουμε το πρωί και το απόγευμα και 12 Ιουλίου μόνο το πρωί. Και πριν να κλείσουμε τη συνεδρία είναι τελευταίο θέμα γιατί είναι ένα θέμα για πολλούς αλλά και για μένα. Είναι σημαντική συνεδρίαση αυτή γιατί θα αποχαιρετήσουμε τον Χεσού Πάρδο που ήταν πολύ αξιόλογος συμμετέχοντας εδώ στην Επιτροπή μας. Θα περάσει σε άλλα καθήκοντα, θα αναλάβει καθήκοντα στη Γεωργία και θα μας εγκαταλείψει και εγώ θα ήθελα ε, να μας εγκαταλείψει έχοντας ε, το γενικό αίσθημα ότι είναι ένα πραγματικά αξιόλογος άνθρωπος και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, σας εύχομαι καλή τύχη για αυτά τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβετε στον τομέα της γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ Χεσούς και καλή τύχη. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Muchas Σας ευχαριστώ όλους. Ο πρόεδρος ευχαριστώ και τους Ευχαριστούμε και εμείς. Πραγματικά εδώ εργαστήκαμε σαν να είμαστε σε αγώνες ράλι.